Κι όμως είμαστε στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2008. Οι συντάξεις ε, περνάνε περίοδο βεβαιότητα. Και αυτό ε, έχει δημιουργήσει προβλήματα και με την εξυπηρέτηση των δανείων ακινήτων των διαφορών οικοκυριών. Έχουμε πτώσεις ε, εκατοντάδων ποσοστιαίων μονάδων, κάποιες περιπτώσεις χιλιάδων. δεν υπάρχει δυνατότητα να εξυπηρετηθούν τα χρέη αυτά. Κάποιοι μπορεί και να οδηγηθούν στη φυλακή ε, επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν τα χρέη του. Και αυτό βεβαίω δημιουργεί καταστροφικέ συνέπειε στην προσωπική ζωή, την υγεία, τι κοινωνικέ συνθήκε των ανθρώπων αυτών. Οι εταιρείε δεν θέλουν να εξυπηρετήσουν του ε, πελάτε του, ούτε οι τράπεζε και οι οικονομικέ δυσχέρειε όλων είναι πολλαπλέ. Εδώ και πολύ καιρό ζητώ καλύτερη προστασία των καταναλωτών για όσου πήραν αυτά τα ε, express δάνεια. Διότι αυτή η επιχειρηματική τουλάχιστον στήματα των τραπεζών πρέπει να απαγορευτεί. Νομίζω θα πετύχουμε μεγάλη ε, στήριξη για κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε ο κύριο Φωζέρ για ένα λεπτό. Κύριε Ντράγκη, θέλω να εκφράσω το θαυμασμό μου. Τι θράσος, τι κότσια είναι αυτά. Με μια οικονομική, δημοσιονομική κρίση που την έχουν προβλέψει όλοι οι εμπειρογνώμονες. Έρχεστε εσείς να μας πείτε ότι όλα πάνε καλά. Θα έπρεπε να το γνωρίζετε και το γνωρίζετε ότι έπρεπε να υπάρχει ομοσπονδιακός προϋπολογισμός για το ευρώ, ενιαίος. Όμως κανείς δεν τον ήθελε αυτόν τον προϋπολογισμό. Εσείς είχατε άλλη επιλογή, άλλη εναλλακτική. Να χρησιμοποιήσετε την κεντρική τράπεζα και να εφαρμόσετε το πρόγραμμα του κυρίου ε, του BPI και ε, όσα έλεγε και η Ιταλία για να χρηματοδοτήσει την πραγματική οικονομία των χωρών του Νότου και να μην υπάρχει τόση ανισότητα. Αυτό δεν το θέλαν το 2012 οι Γερμανοί και σήμερα πώς τις καπουλάρατε με 210, με 2 δις 600 εκατομμύρια δημόσιου χρέους και εξαγορά του. Δημιουργήσατε περισσότερο πλούτο και μεγαλύτερα ελλείμματα. Έχετε αποτύχει. Ευχαριστούμε κύριο Μαριάς για ένα λεπτό. Κύριε Ντράγκη, η ευρωζώνη χρειάζεται άμεσες αλλαγές. απαιτείται κατάργηση του δρακόντιου σύμφωνο σταθερότητας και εγκατάλειψη της λιτότητας και της βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής. η ecd πρέπει να μετατραπεί σε ίστατο δανειστή των κρατών μελών και το ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών τραπεζών πρέπει να αποκεντρωθεί τα κράτη μέλη να ανακτήσουν την νομισματική του κυριαρχία και να μπορούν οι κεντρικέ τράπεζε των κρατών μελών να ασκούν αυτοτελή νομισματική πολιτική μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Η ΕΚΤ πρέπει να πάψει να υπηρετεί τη γερμανική Ευρώπη. Μια Ευρώπη στην οποία η Γερμανία σωρεύει εμπορικά πλεονάσματα και ο Ευρωπαϊκός Νότος αυξημένα ελλείμματα και χρέη. Τέλος, κύριε Ντράγκη, η ΕΚΤ και εσείς προσωπικά οφείλετε να ζητήσετε μια μεγάλη συγνώμη από το φτωχοποιημένο ελληνικό λαό στον οποίο ως τρόικα επιβάλλατε μνημόνια προκειμένου να διασωθούν οι ξένες τράπεζες όπως ομολόγησε άλλωστε και ο ίδιος ο κύριος Ντάισελμπλουμ. Ευχαριστώ. κύριος Φαντάλεν, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, τα τελευταία χρόνια είχαμε 4.000 δισεκατομμύρια τα οποία διοχετεύτηκαν στην οικονομία της Ευρωζώνης. Ένα ποσό μεγαλύτερο από το ΑΕΠ της Γερμανίας. Όλα αυτά σε χώρες ε, όπως η Γαλλία και η Ιταλία που ανέβαλαν για χρόνια τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Και τώρα βεβαίως αντιμετωπίζουν την υψηλή ανεργία και ειδικά ανεργία των νέων. Βεβαίω, ε, εντάξει, ωφελήθηκαν από το φθηνό χτήμα οι τράπεζε, αλλά δυστυχώ οι συντάξει και η αποταμίευση δεν έχουν πλέον κανένα νόημα. Η ΕΚΤ αποδείχτηκε πάρα πολύ ε, ε, ήπια και τελικά το αποτέλεσμα ήταν να μην έχουμε καθόλου οικονομική ανάπτυξη. Θα πρέπει να υπάρξει μεταρρύθμιση όχι προς μία ένωση μεταφορών δημοσιονομικών, αλλά προς μια ένωση που ε, θα είναι πιο ανταγωνιστική. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στη διαδικασία Catch the Έχουμε τον κύριο Μποργέτσιο που έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είναι χιλιάδες οι υποθέσεις ε, παρατυπιών και παρανομιών. Ε, έχει κατηγορηθεί ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενώπιον τη ενιαία αρχή επίλυση διαφορών με τι δραστηριότητε εποπτεία. Η τραπεζική κρίση που ζούμε είναι ένα φαινόμενο, ένα γεγονό που θα πρέπει όλου μα ανησυχεί. Είναι πολύ σοβαρό. Και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σα. Αυτό το θέμα δεν ε, έχει εξεταστεί. Παρόλο που κρούεται ο κόδωνα του κινδύνου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και έχει ε, η επισημάνει τα πλημελήματα ε, τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που βρίσκεται ω ακρογωνιαίο λίθο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Συστήματο και οι τράπεζε τη Ευρώπη κινδυνεύουν να πτωχεύσουν. Είναι σοβαρότατη η ευθύνη ε, για την αξιοπιστία και τη ε, Επιτροπή Επίλυση των Διαφορών, αλλά και για το τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Θα πρέπει κάτι να υποθεί ξεκάθαρα πώς πάνε τα πράγματα. Εμείς εκπροσούμε τους πραγματικούς ανθρώπους, τους πολίτες, το λαό. Γνωρίζουμε πολύ καλύτερα την πραγματική οικονομία που εσείς την τσακίσατε. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Ντομπρόφσκης, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη Πρόεδρε Τράγκη, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, στις εγωικέ μου παρατηρήσεις, αναφέρθηκα στις επικοδηματικές διευθετήσεις και δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πολλές πτυχές της έκθεσης του κυρίου Μάτο μας δείχνουν ότι συνεχίζει να ισχύει αυτό. Παρ' όλα αυτά, στα καταληκτήρια σχολιά μου, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που τονίστηκε και στην έκθεση και αφορά την ανάγκη της ε, οικονομικής ε, ολοκλήρωσης προκειμένου να διευκολύνουμε την ε, υλοποίηση της νομισματικής πολιτικής. Αυτό αφορά την υλοποίηση της ε, Τραπεζικής Ένωσης ε, και την υλοποίηση της Ένωσης Κεφαλαγορών. Η Κομισιόν έχει παρουσιάσει επτά προτάσεις ε, για την Ένωση Κεφαλαγορών. Από αυτές μόνο οι τρεις έχουν υιοθετηθεί και υπάρχει πολιτική συμφωνία για δύο ακόμη. Επομένως, βασιζόμαστε στη συνεχιζόμενη υποστήριξή σας ε, για την Ένωση Κεφαλαγορών που θα οδηγήσει σε καλύτερα συνδεδεμένες κεφαλαγορές ε, και θα ε, προωθήσει και τη διεθνή θέση του ευρώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στον πρόεδρο Μάριο Ντράγκη για να κλείσει τη συζήτησή μας και κατόπιν στον κύριο Μάτο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ και τον εισηγητή, τον κύριο Μάτο, για την έκθεσή σας. Και σας ευχαριστώ όλους ε, για τις φιλοφρονήσεις σας προς την ΕΚΤ. Θα απαντήσω και στις επικρίσεις. Πρώτα απ' όλα για το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων. Το ΕΔΙΣ. Η ΕΚΤ ανέκαθεν υποστήριζε το σύστημα αυτό. Θέλω όμω εδώ να κάνω τρει ε, υποπαρατηρήσει. Πρώτον, όποιο και αν είναι ο δρόμο προ το σύστημα εγγύηση των καταθέσεων, το ΕΝΤΙΣ, ο τελικό στόχο να έχουμε ένα τελικά αντασφαλισμένο σύστημα δεν θα είναι εντό. Δεν θα είναι εύκολο να φτάσουμε ως εκεί. Όλοι το γνωρίζουμε πολλά πισωγυρίσματα, καθυστερήσει, συμβιβαστικέ και διαπραγματεύσει χρειάζονται, είναι απαραίτητε. Όμω η κατεύθυνση έχει οριστεί. Και ορίζοντα των τελικών αποτελεσμάτων είναι μπροστά μα. Το πώ θα αποφασίσουμε να δράσουμε είναι θέμα τη δική σα διακριτική ευχέρεια. Αλλά ό,τι και να αποφασίσετε δεν θα αλλάξει η τελική έκβαση. Και η τρίτη μου παρατήρηση για το ΕΝΤΙΣ είναι ότι δεν υπάρχει σαφής πρόοδος, περίπτωση σαφούς πρόοδου εδώ, εάν δεν υπάρξει μια πιστική μείωση του κινδύνου παντού. Έχουμε ήδη επιτύχει κάποια πρόοδο σε αυτό το μέτωπο, ε, ήδη, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα. Η ΕΚΤ σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλές περιστάσεις, έχει δείξει ότι η κατανομή του κινδύνου από μόνη τη φέρνει μείωση του κινδύνου. Ουσιαστικά δηλαδή ε, οι δύο οδοί αυτές, παράλληλες οδοί αυτής της κοινή πορείας πρέπει να ε, στροφούν ταυτόχρονα. Είναι πολλά τα ερωτήματα που είχαν να κάνουν με τις οικονομικές συνέπειες των πολιτικών της ΕΚΤ. Κάνατε συγκρίσει τη Ευρωζώνη με άλλε περιοχέ του κόσμου, με το τι έγινε πριν την υιοθέτηση του ευρώ, πόσο όμορφο και φανταστικό ήταν ο κόσμο μα πριν το ευρώ. Νομίζω σε μια πρόσφατη ομιλία που εκφώνησα, αλλιώ τα είχα πει εγώ, ιδίω για το πώ ήταν ο κόσμο πριν. Δεν ήταν τόσο φανταστικά τα πράγματα, ιδίω στι χώρε που ο κόσμο παραπονιέται πιο πολύ για το ευρώ. Καθόλου δεν ήταν όλα υπέροχα και όμορφα πριν το ευρώ. Να σα συγκρίνω το τι γίνεται με τη ΣΥΠΑ, γιατί κάποιο το είπε και αυτό το ποσοστό απασχόλησης το 98 στην Ευρωζώνη των 19 ήταν 59,8%. Τώρα είναι 67,3%. Είναι το υψηλότερο που είχαμε καταγράψει ποτέ στην Ευρωζώνη. Στις Ηνωμένε Πολιτείε ήταν 73,9% το 98 και σήμερα είναι ε, 70,6%. Μειώθηκε, δεν αυξήθηκε. Οι θέσει εργασία που δημιουργήθηκαν στην Ευρωζώνη σε αυτό το χρονικό διάστημα είναι 19,8 εκατομμύρια και 17,2 τα εκατομμύρια στα κατημέλη ε, τη Ευρωζώνη. Βεβαίω, οι μονάδε αυτέ πρέπει να ε, ανήκουν στην ενέργεια τη στοιχεία. Και το ίδιο ισχύει και για τα ποσοστά απασχόληση σε εκατομμύρια. Οπότε, όταν με ρωτούν για τις παράπλευρε συνέπειε τη νομισματική μας πολιτική στην ε, Ευρωζώνη, η απάντηση είναι απλή η βασική παράπλευρη συνέπεια μεταξύ του 2013, όταν η κατάσταση ήταν πράγματι χειρότερη για το τι έγινε σήμερα, η πραγματική παράπλευρη συνέπεια ήταν η δημιουργία 9,6 εκατομμυρίων θέσεων εργασία. Περισσότερε από ποτέ. Ε, εδώ ε, κάτι άλλο. Η οικονομική σταθερότητα είναι ε, το τι γίνεται στην κεντρική, στο κεντρικό πυρήνα της Ευρωζώνης και το πόσο οι τιμές ε, πρέπει να πιέζονται μάλλον στην αγορά των ακινήτων και ιδίω σε κάποιες χώρες για την αγορά κινήτων για κατοικίες ή στην αγορά ομολόγων. Όμως αυτό, κάποιος από αυτούς τους κινδύνους μπορεί να δημιουργήσει πραγματικά συστημικά προβλήματα και τριγμούς. Βεβαίω θα παρακολουθούμε όλα αυτά πολύ προσεκτικά. Η απάντηση όμως σε αυτές τις ε, περιορισμένες τοπικά καταστάσεις είναι ότι η νομισματική πολιτική θα πρέπει να συνοδεύεται από την μακροεποπτεία και τις σχετικά εργαλεία που θα πρέπει να ε, ασκούν και να χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα δημοσιονομικά τους εργαλεία σε συντονισμό με την ΕΚΤ. Υπήρχαν και κάποιες γενικότερες ερωτήσεις για το ρόλο της ΕΚΤ και πολύ ορθώς παρατήρησε και ο εισηγητής ότι η ΕΚΤ έχει το ρόλο της αλλά δεν μπορεί να αναλάβει και τα πάντα. Δεν μπορεί να κάνει όσα δεν έκαναν οι υπόλοιποι. Η ΕΚΤ έχει έναν ρόλο που περιορίζεται στην ε, νομισματική πολιτική. Και αυτό ορίζεται ξεκάθαρα στην εντολή τη. Δεν μπορεί να αναλάβει τα καθήκοντα όλων. Υπ' αυτήν την έννοια, Το έχω πει επανειλημμένο και σήμερα το πρωί και όλας. Το θέμα δεν είναι Το θέμα δεν είναι να είχαν όλοι, να, ότι δεν είχαν όλοι τα ίδια ωφέλη. Το πρόβλημα είναι ότι οι χώρε είτε είναι στην Ευρωζώνη είτε όχι, πρέπει να κάνουν μεταρρυθμίσεις. Δεν υπάρχει ένα αποτύπωμα που να είναι πανομοιότυπο για όλους. Ε, το τι πρέπει να κάνει κάθε χώρα αλλάζει ανάλογα με την περίπτωση. Η κάθε μια χώρα έχει τη δική της ιστορία. Αυτό είναι το βασικό. Δεν γίνεται να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς μεταρρυθμίσεις. Και βεβαίω υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Υπάρχουν ελλείψει, υπάρχουν ε, πράγματα που δεν έγιναν στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι κάποια πράγματα που έχουν ήδη αποφασιστεί να ολοκληρωθούν, ιδίω η Τραπεζική Ένωση. Έπειτα είναι να ξεκινήσουμε να προχωρούμε ταχύτερα προς την αγορά την Ένωση Κεφαλαγορών θα πρέπει να δημιουργήσουμε αυτήν την δυνατότητα. Αν γίνουν όμως αυτά τα δύο πρώτα, το Ευρωκοινοβούλιο θα έχει ήδη επιτελέσει με τρόπο θετικό και επικοδομητικό ένα μεγάλο μέρος του ρόλου του. Εάν αυτά τα δύο επιτευθούν, θα τα πάμε πολύ καλύτερα, ακόμη και αν τα επόμενα βήματα για τη δημιουργία της δημοσιονομικής δυνατότητάς μας μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για προφανείς πολιτικούς λόγους. Ε, ρώτησε κάποιος τι μπορεί να κάνει η ΕΚΤ για συγκεκριμένα δάνεια που έχουν ε, δώσει οι τράπεζες τους πολίτες. Γενικώ η ΕΚΤ δεν μπορεί να κάνει και πολλά εδώ. Είναι η αρμόδια εθνική αρχή υπεύθυνη. Πολύ συχνά τα θέματα αυτά είναι θέματα προστασίας του είναι θέματα της Εθνικής Αρχής Προστασίας των Καταναλωτών. Εκείνοι πρέπει να παρακολουθήσουν τους όρους δανειοδότησης. Όμως, ε, γενικώ, εάν υπάρχουν τέτοια εργαλεία σε άλλες χώρες με το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων που κάπου είναι πραγματικά ιδιαίτερα κρίσιμο και δραματικό λόγω των κοινωνικών του συνεπειών, ε, Υπάρχουν δύο περιπτώσεις ε, αυτών που χρωστάνε, δύο κατηγορίες. Μη στρατηγική και αυτή που είναι μέρος ενός ευρύτερου κοινωνικού προβλήματος. Η απάντηση λοιπόν εδώ δεν είναι να αλλάξει απλώς η νοοτροπία των πληρωμών. Περισσότερα πρέπει να βοηθήσουμε τους φτωχότερους. Αυτοί δεν μπορούν να αποπληρώσουν. Θα πρέπει λοιπόν τα δύο πράγματα αυτά να παραμείνουν διαχωρισμένα μην αλλάζετε, μην καταστρέφετε, μην αφοπλίζετε το τραπεζικό σας σύστημα, διότι το αποτέλεσμα θα είναι απλώς να μην μπορούν να δώσουν δάνεια όσο θα ήθελαν στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας της χώρας σας. Βοηθήστε τους φτωχότερους πολίτες που δεν μπορούν να πληρώσουν και να αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Κάτι που ρωτήθηκε από, πολλές, από πολλούς ε, για μια μελλοντική ύφεση. Τι θα γίνει εάν έχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα τα εργαλεία για να τα αντιμετωπίσει αυτά. Η απάντηση είναι πως ναι, έχουμε τα εργαλεία για να απαντήσουμε. Αλλά ας έχουμε υπόψη ότι η τωρινή μας νομισματική ε, θέση είναι ήδη πολύ καλή. Έχουμε αρνητικά ε, επιτόκια. Και αυτό θα κρατήσει μάλλον για αρκετό καιρό. Και παρόλο που έχουμε αποφασίσει να πάυσουμε τις ε, αγορές, τις καθαρές αγορές των περιουσιακών στοιχείων, έχουμε αποφασίσει το επόμενο αποθεματικό να παραμείνει ως έχει για αρκετό καιρό. Δηλαδή όπως τα ομόλογα θα οριμάζουν, θα τα επαναγοράζουμε. Τι σημαίνει αυτό ως προς τα αριθμητικά στοιχεία. Σημαίνει ότι θα συνεχίζουμε να αγοράζουμε σε μεγάλο βαθμό 15 δις αξίας, ομόλογα αξίας 15 δις το μήνα. Δηλαδή χοντρικά αυτό που κάναμε και το προηγούμενο τρίμηνο ή πέρσι. Επίσης, πολλοί περισσότεροι από ένας ρωτήσαν εάν η πολιτική μας έχει βοηθήσει τα αξιόγραφα. Προσπαθήσαμε να λύσουμε εις βάθος τις συνέπειες της νομισματικής μας πολιτικής για την κατανομή εισοδήματο ε, και του πλούτου. Είναι σαφές. Κάθε απόφαση νομισματικής πολιτικής έχει επιπτώσει ω προ την κατανομή. Όταν αλλάζουν τα επιτόκια, αλλάζουμε και το πού πηγαίνει ο πλούτο μεταξύ ε, αυτών που χρωστάνε και αυτού που έχουν δανειστεί, ε, που έχουν δανείσει, των νέων και των ηλικιωμένων. Όμως η ποσοτική χαλάρωση και η αγορά περιουσιακών στοιχείων έχει ορατές συνέπειες, διότι όπως ανεβαίνουν οι τιμές και κυρίως αυτοί που έχουν ε, καλά περιουσιακά στοιχεία είναι πλουσιότεροι, όπως λοιπόν οι τιμές ανεβαίνουν, αλλάζουν τα πράγματα ε, Εάν η πολιτική μα τώρα επιδεινώνει το πώ γίνεται η κατανομή. Εάν δείτε όλε τι συνέπειε μαζί, η απάντηση είναι όχι. Γιατί? Διότι αλήθεια είναι ότι βραχυπρόθεσμα ε, χειροτερεύει ίσω την κατανομή του πλούτου. Όμω, ποια είναι οι χειρότεροι παράγοντε στον παράγοντα ότι επιδεινώνεται η κατανομή περισσότερο από όλου του άλλου παράγοντε. Είναι η ανεργία, το γεγονός ότι η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ είναι επιτυχής αποδεικνύεται επειδή επέτρεψε να έχουμε σαφή ανάπτυξη της απασχόλησης, όπως είπα στην αρχή της παρέμβασής μου. Μία ερώτηση αναφέρθηκε στο σημείο της πρόσβασης των μικρομεσαίων στις πιστώσεις η πολιτική μας έχει εμποδίσει, έχει περιορίσει, έχει οδηγήσει σε συρρήκνωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων στις πιστώσεις. Η απάντηση είναι σε καμία περίπτωση. Το πρόγραμμά μας με τα ομόλογα και το πρόγραμμα της ποσοτικής μας χαλάρωσης επέτρεψε στις ε, τράπεζες και στα ισοζυγιά τους να βρεθεί κι άλλο περιθώριο για δάνεια προς τις μικρομεσαίες. Όλα τα στοιχεία, όλα τα στοιχεία το επαναλαμβάνουν από το 2013 όταν ξεκινήσαμε με τα RTO δεν είναι ε, δάνεια χωρίς όρους. Είναι δάνεια στις τράπεζες υπό τον όρο ότι ε, δανείζουν σε εταιρείε της πραγματικής οικονομίας. Δεν ξέρω εάν αυτό βοηθάει σε τίποτα. για να μιλάμε για έναν κόσμο του παραμυθιούλες και αυτά δεν συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Αλλά κάτι άλλο ενδιαφέρον που προέκυψε από πολλές ερωτήσεις είναι ότι η νομισματική χρηματοδότηση του ελλείμματο είναι η μαγική λύση σε όλα τα προβλήματα. Ε, είχε ερωτηθεί και στο παρελθόν αυτό. Ε, είναι ενδιαφέρον αυτό που υπόθηκε. Διότι όταν υπήρχε η εποπτεία για τις χώρες που ε, χρησιμοποιούσαν τη χρηματοδότηση της εποπτείας πριν το ευρώ, η κατάσταση ήταν πολύ κακή είχαν πολύ ψηλό πληθωρισμό. Είχαν ανεργία υψηλότερη από τις χώρες που δεν είχαν τέτοιου είδους ε, εποπτεία. Εν συντομία λοιπόν αυτό. Αλλά το παράδοξο είναι που ακούμε να προτείνεται αυτή η λύση της ε, χρηματότητας της εποπτείας από ανθρώπους που ήταν κατά, ήταν κατά αυτού ω ε, λε και ήταν το σοβαρότερο έγκλημα, το δεχθέστερο έγκλημα μέχρι χθε. Νομίζω ότι απήντησα στις περισσότερες ερωτήσεις. Μια κουβέντα και για το Outlook. Για το πώς ε, φαντάζει το μέλλον. Ε, εδώ λοιπόν δεν πρέπει να τηρήσουμε ε, στάση ακινησίας. Η κατανάλωση ε, ενισχύεται, οι επενδύσεις επίσης, η στήριξη στους αγοραστές με την νομισματική πολιτική, εξαγωγές λιγότερο. Καλές είναι, όχι και θαυμάσεις. Και η αγορά εργασίας συνεχίζει να είναι εύρωστη. Ωστόσο, όλα αυτά συμβαίνουν με ολοένα και χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. τα δεδομένα που λαμβάνουμε δείχνουν ότι θα έχουμε αυτή την αδυναμία για περισσότερο χρόνο από ό,τι ελπίζαμε πριν από λίγους μήνες. Δηλαδή, ε, στην αρχή είχαμε λιγότερα δεδομένα και λέγαμε και συνεχίζουμε να λέμε ότι αυτός ο ασθενής ρυθμός οφείλεται σε συγκεκριμένους παράγοντες. Ιδίω για στο τι συμβαίνει σε κάποιου τομεί σε κάποιε χώρε, όπω με την αυτοκινητοβιομηχανία στη Γερμανία. Ε, αυτό είναι μια προσωρινή πτώση, α πούμε. Αλλά είπαμε ότι θα υπάρχουν και μονιμότερα αίτια αυτή τη επιβράδυνση. Κάποια από αυτά δεν θα αλλάξουν. Το 2017 είχαμε μια μάλλον ε, μοναδική χρονιά σε σχέση με τους ιστορικούς μέσους όρους μας και περάσαμε σε πορεία χαμηλότερης ανάπτυξης. Όμως η ερώτηση που πρέπει να θέσουμε στους εαυτούς μας είναι Όλο αυτό είναι κάτι το προσωρινό, θα κινηθεί ως σπιράλ ή θα περάσουμε σε μια ύφεση διαρκείας. Περνάμε σε ύφεση γρηγορότερα και για να από ό,τι περιμέναμε πριν. Και πόσο θα κρατήσει αυτή η επιβράδυνση. Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση πρέπει να σκεφτούμε τα γενεσιουργά αίτια αυτής της αποδυνάμωσης της ανάπτυξης και οι παράγοντες αυτοί έχουν να κάνουμε με όσα λέμε καθιστέ, αυτό που έχει συμβεί και στην Κίνα. Δηλαδή με γεωπολιτικές αβεβαιότητες πλέον. Και εδώ, σε εθνικό επίπεδο, μας απασχολεί για πόσο καιρό θα κρατήσουν αυτές οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες. Αυτές θέτουν ένα αμφιβόλο τους πυλώνες επί των οποίων οικοδομήθηκε ολόκληρη η οικονομική μας τάξη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν ε, σωστές επιλογές. Και θα πρέπει βεβαίω να δούμε και πώς ε, προβάλλουν αμφιβολίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λόγω του Brexit, λόγω των όσων έγιναν στην Κίνα, λόγω της απόρριψη του πολυμερούς ε, συστήματος παρατηρούμε ότι κάποια από αυτά τα πράγματα βελτιώνονται και κάποια άλλα χειροτερεύουν. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι τουλάχιστον ε, για το άμεσο μελλοντικό χρονικό διάστημα θα συνεχιστεί η αβεβαιότητα, απλώς θα μεταβάλλεται ε, το είδος της, η φύση της. Αυτό έχει κόστος. Το κόστος είναι η μείωση της εμπιστοσύνης της επιχειρήσης, τους καταναλωτές και γι' αυτό Τώρα αξιολογούμε το πώς ε, διαμορφώνεται η κατάσταση, καθώς ε, σας μιλάω. Πρόεδρε, νομίζω, έχω την εντύπωση, ότι απέντησα στα πάντα. Εάν ξέχασα κανέναν, ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε Τράγκη. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η συζήτηση, το λόγο έχει ο συνάδελφο Μάτο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Ντράγκη, επαναλαμβάνω ότι χαίρομαι ιδιαίτερως για την παρουσία σας, παρόλο που ε, ήταν περισσότερο ομιλία δική σας παρά ανάλυση της ετήσιας έκθεσης του 2017. Παρ' όλα αυτά, ε, χαίρομαι για το, την αναγνώριση που κάνετε το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μακάρι να μηνθούν και άλλοι το παράδειγμά σας. Και ευχαριστώ και τον ε, Αντιπρόεδρο τον Πρόψκη γιατί έκρινε θετικά την έκθεση. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, που έλαβαν μέρος στη συζήτηση, ακόμη και αν διαφωνώ με μερικούς από αυτούς. Συμφωνώ ε, ότι θα πρέπει να είμαστε συγκαταβατικοί και να είμαστε πιο προσαρμοστικοί και να εφοδιαστούμε με μέσα για να αντιμετωπίσουμε νέες κρίσεις. Γιατί έχουμε ήδη την εμπειρία της κρίσης, α μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη. Όντως, η νομισματική μα ένωση είναι πια πιο σταθερή, αλλά υπάρχουν ε, εκρε... εκκρεμότητες, τα κόκκινα δάνεια, το σύστημα εγγύης καταθέσεων. Αυτά τα θέματα θα πρέπει με αποφασιστικότητα να την αντιμετωπίσουμε. Η μείωση και η ε, κοινή ανάληψη κινδύνων θα πρέπει να συμβαδίζουν. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να μην επαναπαυθούμε στις δάφνες μας και να είμαστε φιλόδοξοι και να προχωρήσουμε. Θα ήθελα να σταθώ σε τρία σημεία που έτυχαν σχεδόν αμέριση υποστήριξη των Ευρωβουλευτών. Είναι σημαντικό να βαίνουμε προς μια μεγαλύτερη ε, χρηματοοικονομική σύγκληση με τη ρύθμιση των χρηματομιστών αγορών, ώστε να εξασφαλίσουμε καλύτερη, με περισσότερη σταθερότητα τη Ευρωζώνης. Θα πρέπει επίσης να εκπληρώσουμε τους στόχους της βιωσιμότητας και στο πλαίσιο των νομισματικών πολιτικών. Επίσης ε, και η ΕΚΤ πρέπει να δεσμεύεται από τη Συμφωνία των Παρισίων και θα πρέπει ε, να τηρήσουμε τους στόχους που εγκρίναμε στη Συμφωνία των Παρισίων. Επίσης, κάτι που επισημάνετε και εσείς, το έργο της ΕΚΤ στα θέματα διαφάνειας ήταν πολύ σημαντικό για να βελτιωθεί η ε, προβολή των πολιτικών. Και φυσικά έχετε απόλυτη ανεξαρτησία στην ε, χάραξη τη νομισματικής σας πολιτικής όπως προβλέπετε και από τις συνθήκες. Η λογοδοσία, η μεγαλύτερη διαφάνεια και η ανεξαρτησία είναι τρεις πλευρές ε, του ίδιου τριγώνου και θα πρέπει να ισχύουν και οι τρεις. Σα ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μάτο. Ολοκληρώθηκε εδώ η συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο. Επόμενο σημείο είναι η έκθεση ΤΟΡΒΑΛ σχετικά με την Τραπεζική Ένωση, τη έκθεση για το 2018. Πέντε λεπτά το λόγο έχει ο εισηγητής. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οφείλω να πω πως λυπούμε που βλέπω να αποχωρεί από την αίθουσα ο Μάριο Ντράγκη με το που ξεκινά αυτή η συζήτηση. Γιατί με απογοήτευσε κάπως η προηγούμενη συζήτηση, οφείλω να πω. φαίνεται ότι ορισμένοι συνάδελφοί μου έχουν ξεχάσει τι συνέβη στο παρελθόν. Έχουν ξεχάσει την ιστορία. Τι έγινε κάποιες δεκαετίες πριν, μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο, από το 45 και μετά. Κατά κύριο λόγο, είχαμε μία σειρά σφαλμάτων οικονομικών και υποτιμήσεων, όπως συνέβη με τη Φιλανδία, για παράδειγμα, αλλά και με άλλες χώρες. Και ίσως θυμάστε το 1956 ότι και το Ηνωμένο Βασίλειο είχε αντιμετωπίσει σοβαρέ δυσκολίε. Έκτοτε, τα προβλήματα με τα εθνικά νομίσματα και με τις υποτιμήσεις ε, πολύ απλά συνεχίστηκαν. Ο Βίλι Μπραντ, ε, νέος σοσιαλδημοκράτης, ε, πολιτικός στη Γερμανία, είχε πει κάποια πράγματα τότε. Είχε εκφράσει ανησυχίες για την αδυναμία επίλυσης των οικονομικών προβλημάτων που έβλεπε να αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Τότε είχε προτείνει τα κράτη-μέλη της ε, Ευρώπης να δημιουργήσουν τα προβλήματα με τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Το 20% των αποθεματικών θεωρούσε ότι έπρεπε να δημιουργήσει ένα κοινό αποθεματικό για μελλοντικέ λύσεις. Όμως, γι' αυτό υπήρχε μια προϋπόθεση, ότι έπρεπε να μάθουν οι χώρες να τηρούν τους κανόνες. Και εκεί προέκυψαν και οι δυσκολίες με την πάροδο των ετών. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να ξαναδιαβάσουμε τα λόγια του Βίλι Μπραντ. και να δούμε γιατί μιλά ο Βίλι Μιλά για τα νομίσματα, μιλά για τη Γερμανία, όλος ιδιαιτέρως, και μιλά για τα μέτρα για τη, με τη, τη, σιδηρή, τη σιδηρά γροφιά. Τα οικονομικά μέτρα, τα οποία επαναλαμβάνονται. Από τότε που έλαβε το λόγο ο Βίλι Μπραντ και είπε αυτά, μέχρι σήμερα η νομισματική πολιτική αντιμετωπίζει προβλήματα. Γι' αυτό και δημιουργήσαμε πριν 20 χρόνια το ευρώ. Τώρα έχουμε ένα σύστημα πολύ πιο εύρωστο. Τώρα, κατά πόσον είναι εντελώς προφυλαγμένο και στεγανοποιημένο για να μην πληγεί από κραδασμούς, αυτό που είδαμε το 2008 και το 2009 δείχνει ότι δεν ήταν τόσο ανθεκτικό το σύστημα, ιδίως το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα. Βέβαια έχουν θεσπιστεί κανόνες και όποιοι παρακολουθούν τα τελευταία δέκα χρόνια και κάτι την οικονομική πολιτική θα ξέρουν ότι όταν η Banco Popular της Ισπανίας δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει τι τις πληρωμές της ε, καθαρίστηκε με εφτακτό τρόπο. Η Μπάνκα Κάριτζε ήταν μια άλλη τράπεζα που μπήκε σε διαχείριση από την ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε καθεστώς διαχείρισης. Επομένως, προβλήματα υπάρχουν, έχουμε και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και άλλα προβλήματα. Όμως ε, τώρα είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση σε σχέση με το τι ίσχυε πριν από 50 χρόνια. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ αγαπητέ συνάδελφε Τόρματς. Εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το λόγο τώρα έχει ο επίτροπο κύριος Ντομπρόμσκης. Uh, Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, Καταρχά να ευχαριστήσω τον κύριο Νίλ Τόρβαλτ για την ετήσια έκθεσή του για την Τραπεζική Ένωση. Η έκθεση μα δίνει έξοχο απολογισμό σχετικά με το πώ τα Πεζική Ένωση πρόθεσε νέα αγορά, συνήβαλε στου θεμητού όρου του ανταγωνισμού και στη χρηματοστατική σταθερότητα. Πολλά έχουν επιτευχθεί από τον αρχικό σχεδιασμό όσον αφορά το ρυθμιστικό και υποπτικό πλαίσιο για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο ακόμα. Η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ενώσεως είναι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και καλωσορίζουμε το ότι υπογραμμίζει έκθεση στη συνεχή προσπάθεια προς επίτευξη των λόγων στόχων. Από την περσινή συζήτηση, πρέπει να πω, στο χρόνο που πέρασε είχαμε απτή πρόοδο. Καταρχάς, έχουμε συμφωνία επί του τραπεζικού πακέτου, όπως αποκαλείται, ο Γκούνερ Χόκμαρ και ο Πέτερ Σίμον το διαπραγματεύτηκαν αυτό, εκ μέρους του Κοινοβουλίου. Το τραπεζικό αυτό πακέτο θα ενισχύσει το πλαίσιο συνετής ε, διαχείρισης ε, προληπτικών μέτρων και θα αντιμετωπιστούν καλύτερα οι κρίσεις χωρίς να χρησιμοποιούνται τα χρήματα των φορολογωμένων. Τεχνικό έργο για ολοκλήρωση αυτού συνεχίζεται και προσβλέπουμε σε έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου, ούτως ώστε το Κοινοβούλιο να ολοκληρώσει το έργο του πριν τις διακοπές των εργασιών Δεύτερον, σημαντική πρόοδο επετέφθη όσον αφορά την εφαρμογή του σχεδίου δράσεω που θετήθηκε από το Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2017 για τη μετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δάνειων και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σειρά ανακοινώσεων και προτάσεων πάνω σε αυτό. Και ε, έχουμε επίσης ε, έχουμε και συμφωνία για το μέτρο ασφαλείας για να μην σωρεύονται στο μέλλον μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Πρόσφατα έχουμε δει το 2018 τα κεφα... τα κεφ... η θέση κεφαλαίων των τραπεζών έχει ε, βελτιωθεί, η δανειοδότηση των τραπεζών έχει μειωθεί και οι δυνατότητες έχουν αυξηθεί. Ταυτόχρονα τα κόκκινα δάνεια εξακολουθούν να μειώνται οι τράπεζες και έχουν δημιουργηθεί και τα σχετικά αποθέματα απορρόφησης κραδασμών. Ενθαρρύνεται ε, διότι βλέπει ότι έχουν μειωθεί τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε διάφορα κράτη-μέλη, κυρίως μέσω των δραστηριοτήτων των διαφόρων φορέων και των τραπεζών. Έχουμε διαφορετικά επίπεδα μη εξυπηρετωμένων δανείων στα διάφορα κράτη-μέλη. Πρέπει να, η διαφορά αυτή να καλυφθεί και αντιμετωπιστεί και το σχέδιο δράσεω για αυτά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια πρέπει να εφαρμοστεί πλήρω. Τρίτον, διάφορα σκάνδαλα ξεπλήματο χρήματο, τα οποία μπλέκονται στι ευρωπαϊκέ, ε, ανεφάνισαν το 2018 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε νομοθετικού περιεχομένου προτάσει σχετικά με αυτό και συνοδευτικές ε, ανακοινώσεις για την ενίσχυση του πλαισίου της ενώσεως για την καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος, σχετική εποπτεία και τα προληπτικά μέτρα. Έχουμε βρει πακέτο μέτρων που θα ενισχύσει τις τρεις εποπτικές ευρωπαϊκές αρχές και τα εργαλεία που διαθέτουν όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων και ορίζω τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου που υθέτησε μόλι τώρα βάσει της εκδόσεως της Περβάνς περέ και του Οκμαρτ Κάρα και βασίζομαι στην πλήρη υποστήριξή σα για να ολοκληρωθούν διαπραγματεύσει όσον αφορά προτάσει νομοθετικού περιεχομένου πριν το τέλο τη παρούση θητεία. Η έκθεση ε, των τραπεζών σε κρατικά χρέη. Εκεί έχουμε ήδη άποψη με το Κοινοβούλιο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχει σοβαρό αντιχτυπώ. Το 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε προτάσει για αριθμιστικό πλαίσιο για, τα αξιόγραφα αυτά τα κρατικά και να μειωθεί οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων ε, κρατικών ομολόγων και των τραπεζών. Όσον αφορά το Fintech, χρειάζεται να έχουμε ισότιμους όρους ε, ανταγωνισμού μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά και θα πρέπει να συμμετέχουν οι νέες καινοτόμες τεχνολογίες στον χρηματοστικό τομέα. Αυτό είναι κάτι το οποίο αντικατοπτρίζει στην ανακοίνωσή μα για το FinTech, που είχε τη μορφή σχεδίου δράση και κάλυψε διάφορε πρωτοβουλίε για την ενίσχυση μεταξύ άλλων και την αντοχή σε κυβερνοεπιθέσει. Όπως ανέφερα, παρά όλα τα βήματα προόδου, ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο στόχο. Πρέπει να γίνουν περισσότερο όσον αφορά το κοινό μέτρο ασφαλείας για το κοινό ταμείο ρευστοποίηση και το σύστημα εγγύησεως καταθέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ίδις αναγνώρισε η έκθεση τη σημασία συνεχιζόμενων εργασιών από αυτών των προτάσεων όσον αφορά το κοινό αυτό δίχτυ ασφαλείας, το backstop. Προδεύουμε η συμφωνία του Δεκεμβρίου του 2018 στην Σύνοδο Κορυφή για το ευρώ θα πρέπει να εφαρμοστεί τάχιστα και να μπει στην αλλαγή συνθήκη του ESM, ελπίζουμε μέχρι τα μέσα του νεστότο έτου και θα πρέπει να προχωρήσουμε με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα που θα παρέχει ένα δίκτυο ασφαλεία και αυτό θα πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο το ενωσιακό. Θα διευρύνει διευρυνθεί έτσι ο δημοκρατικό έλεγχο των δραστηριοτήτων αυτού. Δυστυχώ δεν έχουμε προχωρήσει τόσο όσον αφορά τη δημιουργία του EDIS που βασικά είναι ο τίτλο πυλώνα τη Τραπεζική Ενώσεω. Σα παροτρύνω λοιπόν να ολοκληρώσετε την έκθεση υπό την ηγεσία του κ. Έστερ Ντελάγκερ σε αυτή τη θητεία για να δείξουμε το Κοινοβούλιο που στηρίζει αυτή την προσπάθεια και σα παροτρύνω να εξετάζετε την Τραπεζική Ένωση και να την θεωρήσετε σαν πρωτοβουλία που είναι υποφελή για όλου του Ευρωπαίου. Έχουμε πετύχει πολλά μετά από το ξέσπασμα τη κρίσεω, πραγματικό θετικό αντίκτυπο είχαμε για τι επιχειρήσει και τα νοικοκυριά με τα μέτρα μα. Ταυτόχρονα θα λογοδοτήσουμε για τον κίνδυνο που δημιουργείται από μια τελή Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, θα πρέπει αποτελεσματικά να χρησιμοποιήσουμε τον υπολοιπόμενο χρόνο σε αυτό το πολιτικό κύκλο για να σημειώσουμε την πρόοδο προς την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε Ντομπρόφσκης. Ενάμιση λεπτό το λόγο κύριος Χέκμαρκ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε τον ε, εισηγητή μα και ευχαριστώ και τον Επιτρόπο τον Πρόφσκης. Σήμερα το πρωί εορτάσαμε την 20η επέτειο του ευρώ, του ενιαίου νομίσματος και διαπιστώσαμε πόσο αλλα... πόσες αλλαγές έγιναν ακόμη και πρόσφατα. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές αναλύουν περισσότερο τους κινδύνους, αναλαμβάνουν κινδύνους και κατανέμουν τους κινδύνους και με τα διάφορα βήματα που κάναμε και με βάση τους ακρογωνιαίους λίθους της Ταπεζικής Ένωσης που θέσαμε, σήμερα έχουμε καλύτερη ευκαιρία για την ανάλυση των κινδύνων. Και αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτήματα που μας έδωσε ο κανονισμός, η οδηγία μάλλον για την ανάκαμψη και εξυγίαση ε, τραπεζών. Αλλά και η ίδρυση, η θέσπιση των εποπτικών αρχών είναι σημαντικό. Επίσης, πάντα θα έχουμε κρίσεις. Το θέμα είναι πώς θα τις αντιμετωπίζουμε. Πόσο καλά θα τις αντιμετωπίζουμε και πόσο εύκολα θα εξερχόμαστε από τις κρίσεις. Και μάλιστα η θέσπιση του μηχανισμού προστασίας, του backstop, αλλά και η καλύτερη νομοθεσία που ελπίζω να εγκρίνουμε για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα είναι ε, τμήμα αυτής της ε, ρύθμισης και σίγουρα θα πρέπει ε, να ενημερώνονται οι καταθέτες ότι από τη στιγμή που επενδύουν στις τράπεζες αναλαμβάνουν και αυτή κίνδυνο. Επίσης, με τη, την οδηγία για την ανάκαψη και εξήγηση τραπεζών και με το, την οδηγία για τις κεφαλαϊκές απαιτήσει έχουμε πολύ καλύτερες προϋποθέσεις για να αντιμετωπίσουμε τις ε, επερχόμενες κρίσεις και να εξέλθουμε πιο αλόβητοι από ό,τι στο παρελθόν ή με λιγότερα τραύματα από ό,τι στο παρελθόν. Και ευχαριστώ τον εισηγητή και τον Επίτροπο, γιατί σίγουρα έχουμε ακόμη μακρύ δρόμο μπροστά μας, αλλά θα πρέπει να υποτιμούμε τα μέχρι τώρα επιτεύγματά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χέκμαρκ. Ο κύριος Φερνάντες για 1,5 λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ και καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν που είναι εδώ. Καταρχά, φυσικά και οφείλω να ευχαριστήσω τον Νίλ Τόρβαλ, τον εισηγητή τη έκθεση, ε, για το πνεύμα συνεργασία που επέδειξε, όπω και όλου του εισηγητέ, ε, γιατί προσπαθήσαμε από κοινού να καταλήξουμε σε αυτό το κείμενο, ε, συνεργατικό κείμενο που θα ψηφίσουμε αύριο. Θα ήθελα να πω πάντω ότι σε αυτέ τι εκθέσει, όπου και αξιολογούμε τη λειτουργία τη Τραπεζική Ένωση, ενώ είναι σκόπιμε και χρήσιμε, αυτό που είναι σημαντικό για αυτέ είναι να μπορέσουμε επιτέλους να συμπληρώσουμε το θεσμικό πλαίσιο της Τραπεζικής Ένωσης. Το κοινοβούλιο αυτό κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες αυτή τη θητεία, ιδίω δε τους τελευταίους μήνες, για να δει τη δέσμη μέτρων για την απομίωση των κινδύνων, τραπεζική δέσμη μέτρων, ε, για ε, τις ε, εντάξει, μη εξυπηρετούμενα δάνεια κτλ. Χρειαζόμαστε και μια πρόσθετη προσπάθεια όμως τελευταίους μήνες που έρχονται για να μπορέσουμε να έχουμε και την εγγύηση των καταθέσεων για το σύνολο της Τραπεζικής Ένωσης. Ε, έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε ε, ένα προϊόν για την τιτλοποίηση του δημόσιου χρέους ε, που ουσιαστικά θα είναι ένα ασφαλές δημόσιο ομόλογο και θα είναι και ένας μηχανισμός ασφαλείας, ένα backstop που θα στηρίζει αυτό το Ταμείο Εξυγίανση. Έχουμε κάνει βήματα, όπω είπα, για την μείωση των κινδύνων. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και άλλα βήματα που πρέπει να γίνουν και γι' αυτό ζητώ, τολμώ να ζητήσω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δείξουμε τη δυνατότητα αυτού του μήνε να του εκμεταλλευτούμε, να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε για να ε, ολοκληρωθεί και αυτό το σύστημα εγγύηση καταθέσεων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη λειτουργία τη Τραπεζική Ένωση και για την αποφυγή κρίσεων σαν αυτέ που βιώσαμε την τελευταία δεκαετία. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Φερνάντεθ. Επόμενο για ένα λεπτό είναι ο κύριο Έζεκ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ τον εισηγητή για την πολύ ισορροπημένη ε, έκθεσή του που περιέλαβε και τις απόψεις όλων των πολιτικών παρατάξεων. Σίγουρα θα πρέπει να περιορίσουμε το κίνδυνο, ενώ ταυτόχρονα να αυξήσουμε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Χαίρομαι που στην έκθεση Τόρβαλτς ε, λαμβάνεται υπόψη η ποικιλομορφία των διαφορετικών τραπεζικών μοντέλων και ε, η αναγνώριση του ενιαίου συστήματος. Επίσης, πολύ σωστά ο εισηγητής ε, μιλά για την ανάγκη καταπολέμησης ε, της νομοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και του περιορισμού των κόκκινων δανείων και των διαστάσεων της χειόδους τραπεζικής, που είναι περίπου το 40% του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος, όπως υπολογίζεται σε πρόσφατη έκθεση. Η πολωνική αντιπροσωπεία του κόμματο ε, των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών θα υπερψηφίσει την έκθεση Τόρβαλτ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Οζούκ. Κύριο Βιέγα, επόμενο ομιλητή. Σα ευχαριστώ. Το θέμα που καλούμαστε να θέσουμε εδώ είναι έχουμε ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα ικανό να επιλύσει τα προβλήματα της οικονομίας. Η αλήθεια είναι ότι το ίδιο χρηματοπιστωτικό σύστημα εξακολουθεί να είναι το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντί να είναι η λύση. Και ακόμα προβληματίζει η ενάργεια των στοιχείων του ενεργητικού της τράπεζας. Αλλά τι γίνεται με τους μηχανισμούς που ήταν η αιτία αυτού του κερδοσκοπικού ε, φαύλου κύκλου που ήταν η αιτία του χρημα, της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Είχαμε ένα απλό καλοπισμό μετά την Τρίτη Συμφωνία της Βασιλείας ε, με κάποιες ρυθμίσεις ε, για τις τράπεζες, αλλά έχουμε, ε, εξακολουθούμε να έχουμε μεγάλο ποσοστό κόκκινων δανείων και επίσης τράπεζες μεγαθύρια που θα συνεχίσουν να μας δημιουργούν τεράστια προβλήματα στο μέλλον λόγω του συστημικού τους χαρακτήρα θα πρέπει το, το Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας να τεθεί στο, στην υπηρεσία του Ταμείου Εξυγίασης και Ανάκαμψης των Τραπεζών, δηλαδή περισσότερα δημόσια κονδύλια ε, και καλύτερος ε, έλεγχος του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ώστε οι τράπεζες να εξυπηρετούν την οικονομία, όχι το συμφέρον τους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μονό για ένα λεπτό. Ε, κύριε Πρόεδρε, για του Γάλλου πατριώτε, η οδηγία, η φεδεραστική τη Τραπεζική Ένωση είναι νομοθεσία πολιταρχική και αντιδημοκρατική απολυταρχική, διότι από το 1994 χάσανε τραπεζική του κυριαρχία υπέρ τη ε, Ευρωπαϊκή Κεντρικής Τράπεζα. Είναι υπερεθνικό φορέας, ανεξάρτητο από κάθε κράτο και δεν υπόκειται σε κανένα δημοκρατικό έλεγχο στην πραγματικότητα. Μεταφορά των εξουσιών στου τεχνοκράτε που δεν έχουν εκλεγεί τη Φραγκφούρτη, οι εθνικοί μα ηγέτε διέπραξαν σοβαρό σφάλμα να αποκόψουν τον οργανικό δεσμό μεταξύ κράτου και τραπεζικού συστήματο. κάτι που καθιστά τα κράτη εντελώ αδύναμα. Στην επόμενο συστημικό κλειδονισμό και στο μεγάλο κράχ των χρηματιστικών αγορών, οι καταθέσεις στις τράπεζες ε, θα ε, λαφυραγωγηθούν των καταθετών. Λοιπόν, εκτίθουν, ε, οι χρηματοπιστωτικοί φορεί μονίμω εκτίθεται σε κινδύνου και η οδηγία φεδελαστική τη Τραπεζική Ένωση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για την κοινωνικονομική ευστάθεια των κρατών τη Ευρωπαϊκή Ενώση. Ονόμα τη Δημοκρατία και του κοινού ωφέλου των πολιτών θα πρέπει να δεθεί κατεπηγόντω τέρμα σε αυτή την διαστρέβλωση την ευρωπαϊστική τη Τραπεζική Ένωση και θα πρέπει τα κράτη-μέλη σε εθνικό επίπεδο να τον έχουν των τραπεζών του, άρα και οι λαοί να ελέγχουν τι τράπεζε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Μόνο. 1,5 λεπτό τώρα έχει το λόγο ο κύριος Λάγκεν. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή διότι σε μεγάλο βαθμό ε, δέχθηκε τη θέση του ΕΛΚ. Είναι καλή έκθεση αυτή. Ακούσαμε τους δύο τελευταίους ομιλητές, εκπρόσωπο της ΓΚΟΕΑ και εκπρόσωπο του FTD. Έχουμε τις τροπολογίες τους. Θέλει διάλυση της Τραπεζικής Ένωσης η ΓΚΟΕ και η FTD ε, θέλει για την Ιταλία να μπορεί να ε, κάνει κάτι αυτόνομο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και να ποια είναι τα σημαντικά για εμάς σημεία. Όλοι γνωρίζουμε ότι ε, η τραπεζική κρίση ε, οδήγησε, ε, μάλλον προκλήθηκε από την έλλειψη ρυθμίσεων. Υπήρχε μεγάλη απληστία επίση στον κλάδο αυτό. Υπάρχουν λοιπόν σε αυτές οι προτάσεις και χαίρομαι που έχουν κατατεθεί, ελπίζουμε να εφαρμοστούν. Αυτό το οποίο θεωρούμε σημαντικό καταρχάς είναι η αναλογικότητα μεταξύ και μεγάλων τραπεζών στην Αμερική, για τη Wall Street ε, και για τη Main Street υπάρχουν ρυθμίσει για του μεγάλου και για του μικρού. Δεύτερον, αγώνα κατά της νομοποίηση προσώπων από παράνομε δραστηριότητε. Θα πετύχει μόνο αν εφαρμοστούν τα μέτρα από τα κρατημέλη. Τρίτον, ε, το, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα πρέπει ε, να αποσυντεθούν. Και το τέταρτο, αυτό το μοντέλο που υπάρχει δεν θα πρέπει να τεθεί υπό αμφισβήτηση. έχουμε το παράδειγμα τη Γερμανία που το προσπαθεί. Και το τελευταίο είναι το σύστημα σύστημα των καταθέσεων που αυτό θα πρέπει ε, να είναι το πρώτο αν θέλουμε να μειώσουμε τους κινδύνους ε, και ελπίζω να το πετύχουμε μέχρι το τέλος της θητείας ε, στην επόμενη. Επόμενος ομιλητής η κυρία Μπερές για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρο, εξετάζουμε μία πολύ χρήσιμη έκθεση για την κατάσταση της Τραπεζικής Ένωσης. Μας υπενθυμίσατε διάφορα σημεία. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω πως η καλή λειτουργία, η εύρυθμη λειτουργία της Τραπεζικής Ένωσης είναι απολύτως απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία ολόκληρης της οικονομίας. Και θα ήθελα να σταθώ κυρίως σε δύο μηνύματα. Το πρώτο είναι ότι θα πρέπει να είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι, να πάμε ακόμη πιο μακριά. Αναφερθήκατε στην καταπολέμηση της νομοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Και γι' αυτό θα πρέπει να ενισχύσουμε την αρχή, και αυτή ήταν η επιλογή σας και σας στήριξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, ώστε μαζί με τις άλλες εποπτικές αρχές ε, να πρωτοστατήσουν στην καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος ε, και θα είναι αποφαστική η συμβολή τους. Επίσης θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τη διακυβέρνηση των εποπτικών αρχών και θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει στην εντολή που δώσαμε με μεγάλη πλειοψηφία στην αρμόδια επιτροπή. Το δεύτερο μήνυμα που θα ήθελα να διατυπώσω είναι η περίφημη αυτή συζήτηση μεταξύ μείωση και επιμερισμού των κινδύνων. Έχουμε την αίσθηση ότι κάποιοι ευρωβουλευτέ ή κάποια κράτη-μέλη έχουν την ικανότητα μιας σταδιακής ολίσθησης των απαιτήσεων με απαράδεκτο τρόπο. Ε, το ΕΝΤΙΣ, αυτό το σύστημα ασφάλισης καταθέσεων, είναι τμήμα της ε, Τραπεζικής Ένωσης από την πρώτη μέρα θέσπισης. Οπότε, ό,τι κάναμε για τη μείωση των κινδύνων υπό την πίεση του χρόνου με έτοιμα των κρατών μελών, θα πρέπει να συνοδεύεται, θα πρέπει να συμβαδίζει και να αντισταθμίζεται με κάποιο τρόπο από αυτό που ήδη οφείλουμε την δέσμευσή μα υπέρ του ΕΝΤΙΣ, του Ευρωπαϊκού Συστήματο Ασφάλιση Καταθέσεων. Ε, και γι' αυτό προσβλέπουμε και εδώ στην πυγμή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για να σημειώσουμε πρώτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ένα λεπτό τώρα κύριο Σταρμπάτη. Κύριε Πρόεδρε, είπαμε με τον Μάριο Ντράκη πριν ένα χρόνο εδώ ότι το σε αυτό το σύστημα εγγύηση των καταθέσεων, είναι ένα σημαντικό κομμάτι τη Τραπεζική Ένωση. Το είπε και ο Φορνάντε, το είπε και ο κύριο Λάγκεν, μίλησε για τη μείωση κινδύνων. Πράγματι, αυτό ο μηχανισμό εγγύηση των καταθέσεων ε, θέλουμε να κάνει την Ένωση πιο ε, ασφαλή. Την κάνει όμω πιο ανασφαλή, γιατί βλέπουμε τι γίνεται με τι ε, τράπεζε που κάνουν διάφορες διάφορα ρετουσαρίσματα στους ισολογισμούς τους. Ε, έπειτα έχουμε αυτά τα κακά δάνεια, τα κόκκινα δάνεια ε, που τα έχουν οι τράπεζες ε, και αυτό δεν θα το έκαναν. Και έχουμε και τον ηθικό κίνδυνο γιατί τελικά αν, είναι όλοι, αν έχουν όλοι ευθύνη δεν έχει κανένας Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε πιο ασφαλή την Ένωση για να αποφύγουμε την επιμόλυνση, τη μετάδοση κινδύνων από τη μια στην άλλη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ουρμπάν Κρέσπο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάνε 11 χρόνια από τότε που ξεκίνησε η χρηματοπιστωτική κρίση και με η ρηξικέλευτη μεταρρύθμιση του τραπεζικού συστήματο που είχατε αναγγείλει έχει αποτύχει παταγωδό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα δεν είναι καλύτερα προστατευμένη απέναντι σε μελλοντική χρηματοπιστωτική κρίση. Η Τραπεζική Ένωση προωθεί μια όλο και μεγαλύτερη συγκέντρωση στο κλάδο. Ενώ οι μικρομεσαίες τράπεζες γίνονται έρμεο των μεγάλων και τις καταβροχθίζουν οι μεγάλες. Ουσιαστικά προωθείται ένα ολιγοπόλιο που ε, δεν εγγυάται καμία τράπεζα να μην διασωθεί με δημόσια κονδύλια. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πιέζει, πιέζεται να, ε, να, να διαθέσει τα λιγότερα ε, εξασφαλισμένα στοιχεία του ενεργητικού, γίνοντας έρμεο στα ταμεία όρνια. Χρειαζόμαστε ένα σταθερό χρηματοπιστωτικό σύστημα υπό ε, λαϊκό και δημοκρατικό έλεγχο. Δυστυχώ, η Τραπεζική Ένωση μα οδηγεί προ τελείω αντίθετη κατεύθυνση. Δεν είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Ε, αντίθετα, συνεχίζουμε να προσπίζουμε τι τράπεζε ει βάρο των ανθρώπων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Ορμπάν Κρέσπο. Ένα λεπτό, ο συνάδελφο Βάλι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λυπούμε που ο συνάδελφο Λάγκερ αναχώρησε αλλά είπαμε ότι θέλει, είπε ότι η ομάδα μα θέλει να βοηθήσει τι Ιταλικέ τράπεζε και αυτό θέλει να βοηθήσει τι Γερμανικέ τράπεζε. Θέλω να όλο ποιε είναι οι σκέψει του για την Nordbank, όπου είναι πολύ εκτεθειμένη σε, στον τομέα τον ναυπηγικό και στον ναυτιλιακό. Ίσως θα πρέπει να λάβει υπόψη μια κάποια ευαίσθητη τοποθέτηση όσον αφορά τα μεγάλα αποθέματα των μη εξυπηρετούμενων δάνειων. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τον έλεγχο που ασκεί ε, παίρνει κάποιες, ακούει κάποιες συστάσεις από ιδιωτικές τράπεζες. Το είδαμε στον τύπο και στη Γερμανία, από την BlackRock, στην αξιολόγηση που έγινε στις ε, δοκιμές αντοχής και θα μπορούσε να δείξει μεγαλύτερη ευαισθησία όσον αφορά ένα θέμα αυτού του είδους. Η Γερμανία, η Γαλλία, έχουν λάβει εκατοντάδε ε, δισεκατομμύρια ευρώ για να σώσουν τράπεζε του. Η Ιταλία καταβάλει μεγάλε προσπάθειε και έχει μειώσει πάρα πολύ ε, τα μία ε, εξυπηρετούμενα δάνεια και θα πρέπει να υπάρξει κάποια ευαισθησία και σεβασμό για εκείνου που αυτή τη φάση κάνουν προσπάθειε για να αποφύγουν να δημιουργηθούν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα και για τη χώρα και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε, Ευχαριστούμε, Το λόγο έχει για 1,5 λεπτό κύριο Ροζάτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμφωνώ ότι κάναμε σημαντική πρόοδο στη δημιουργία της Τραπεζικής Ένωσης, αλλά πάνε περίπου 7 χρόνια. Και σίγουρα είναι η μητελέ το οικοδόμημά μα αυτό τη τραπεζική Ένωση. Θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη τρία στοιχεία που κατά την γνώμη μου έχουν κεφαλαιώδη σημασία για να λειτουργήσει στο έπακρο και εύρυθμα η Τραπεζική Ένωση. Καταρχήν θα πρέπει να ολοκληρώσουμε το σύστημα, τη διαδικασία της ε, χρηματοδότησης ε, για τη, του Ταμείου Ανάκαμψης και Εξηγήσεων των Τραπεζών. Εδώ και χρόνια ασχολούμαστε με το θέμα της μεταμόρφωσης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας σε αυτό το μηχανισμό για την ανάκαμψη και την εξηγήση των τραπεζών. Επίσης, ακόμη περιμένουμε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων, πολύ απαραίτητο στοιχείο της Τραπεζικής Ένωσης. Και τρίτον, δεν πρόκειται ε, να ε, τα βγάλουμε πέρα με το μεγάλο αριθμό των κόκκινων δανείων. Είναι ένα τεράστιο βάρος που μπορεί να μας δυσκολέψει πάρα πολύ την έξοδο από την κρίση. Κύριε Πρόεδρε, 1,5 λεπτό δικαιούμε. 1,5 λεπτό δικαιούμε, όχι ένα. Λοιπόν, ο μεγάλος αριθμός των κόκκινων δανείων μπορεί να μας ε, δυσχεράνει την έξοδο από την κρίση ή να επιταχύνει την επόμενη ύφεση. Θα πρέπει λοιπόν να επισπεύσουμε τις διαδικασίες προκειμένου να διεκπαιρεώσουμε την Τραπεζική Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ροζάτη. Ναι, συγγνώμη, ε, ήταν λάθος μου. Επόμενη για 1,5 λεπτό κυρία Πιετικάινεν. Ευχαριστώ πολύ. Δέκα χρόνια μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση είναι μια καλή στιγμή να δούμε τι συνέβη και πώς ε, αντιμετώπισαν τα προβλήματα οι θεσμοί μέσω της Τραπεζικής Ένωσης. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί έθεσε όλες αυτές ε, τις προϋποθέσεις για την ίδρυση της Τραπεζικής Ένωσης ήδη από αυτήν την θητεία. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω για την κατανόηση που δείξει σε πολιτικό επίπεδο. Τώρα υπάρχουν τρία ζητήματα. Η υπερχρέωση εξυπηρέτηση του χρέους, ε, οι επενδύσεις ε, με μεγάλο ε, ρίσκο Ήταν κάποια θέματα τα οποία δεν λύθηκαν, εκκρεμούν. Έχουμε και τη βιώσιμη χρηματοδότηση, φυσικά, τις τραπεζικές συναλλαγές, τις δανειοδοτήσεις κτλ. Αλλά και ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η ρύθμιση άλλων ε, ταμείων πιο αρπακτικών επιθετικών, όπως τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου ή άλλα, ώστε οι μικροί επενδυτές να μην ξανααντιμετωπίσουν τους ίδιους κινδύνους που αντιμετώπισαν ε, με τον τραπεζικό κλάδο. Και το Κοινοβούλιο και, το, ε, και η Επιτροπή θα πρέπει να βρουν λύση σε αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε την κυρία Πιετικά. Να περνάμε στη δικασία προσέλκυση τη προσοχή του Προέδρου. Ο κύριο Καπούτο είναι ο πρώτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξασφαλίσουμε σταθερότητα τη χρηματοπιστωτική που χρειάζεται να ολοκληρώσουμε την Τραπεζική Ένωση υιοθετώντα μέτρα που θα μειώσουν τον τραπεζικό κίνδυνο. Στόχο τη Τραπεζική Ενώσεω είναι να εγγυηθεί τη χρηματοδοτική σταθερότητα αλλά και να διατηρήσει την ποικιλομορφία των βιωσίμων τραπεζικών μοντέλων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, αποφεύγοντα να οδηγήσουν το τραπεζικό το σύστημα προ ένα μοντέλο ενιαίο που θα είναι κάτι που θα είναι κακό για τις μικρές τράπεζες. Διότι τέτοια ποικιλομορφία επιτρέπει να καλύψουμε καλύτερα τις απαιτήσει ε, των πολιτών τους και των εγχειρημάτων τους. Θα πρέπει να φροντίσουμε την ευρωπαϊκή εποπτεία. Χρειάζεται προσέγγιση κοινή τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω όσον αφορά ε, την καταπολέμηση του ξεπλήματο χρήματο μέσω τραπεζών. Θα πρέπει σαφώ να καθορίζονται οι διάφορε αρμοδιότητε και να καθορίζεται η αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Δεν κρύβουμε τι ανησυχίε που υπάρχουν τη διάδοση του τραπεζικού συστήματο του Σκιώδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι περίπου 40% του χρηματοστικού